Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καθίσουν. Έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επομένως, ε, ε, να σας πω δύο λόγια για την διοργάνωση των εργασιών μας σήμερα το πρωί. Θα θυμάστε ότι μέχρι τις 10 γίνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Τάξη. Εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης των Ελίζα Φερέιρερ και Τόιερ μαζί με τους σκιώδες εισηγητές. Τους καλημερίζω. Συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και σήμερα είναι χρήσιμο να δούμε ποιες ήταν οι εξελίξεις, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πόσο έχουν προχωρήσει οι κοινέ τους εργασίες συνεισηγητών και σκιωδών εισηγητών. Το νέο στοιχείο συγκριτικά με αυτά που αποφασίσαμε την περασμένη εβδομάδα είναι η απόφαση που ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων και επιβεβαιώθηκε από ψηφοφορία στην Ολομέλεια χθες να οργανώσουμε επί τη ευκαιρία της μίνι συνόδου στις 10 Μία ψηφοφορία που είναι σημαντική για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αναφορικά με την μεταναστευτική κρίση. Συμφωνήθηκε ε, με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του Προέδρου Γκουαλτιέρη και του Προέδρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι στις 10 θα αναστείλουμε ε, θα διακόψουμε τις εργασίες μας για ένα τέταρτο, θα διασχίσουμε το διάδρομο που βρίσκεται απ' έξω για να πάμε στην Ολομέλεια για να ψηφίσουμε τάχιστα το τελικό κείμενο με πολύ λίγες τροπολογίες και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να ξεκινήσει η ακρόαση του Προέδρου Γιούνκερ και του Επιτρόπου Μοσκοβισή στις 10 και 4, αντί για τις 10 που είχε προβλεφθεί αρχικά. Ελπίζω ότι μπορώ να πείσω τους προσκεκλημένους μας να παρατείνουν για ένα τέταρτο την παραμονή τους εδώ στην Επιτροπή μας, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να εξαντλήσουμε ε, την μία και μισή ώρα που έχουμε και έχουν συμφωνήσει να συναντηθούμε. Στη συνέχεια λοιπόν στις 10 και 4 θα είναι κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οίκων και Τάξ. Και στη συνέχεια πάλι σε κοινή συνεδρίαση Οίκων και Τάξ των δύο Επιτροπών θα ε, δούμε την Επίτροπο Φεστάγκερ και ελπίζω και εκείνη να την πείσουμε να παρατείνει την παρουσία της εδώ κατά ένα τέταρτο αφού η δική της ακρόαση και η συνάντησή μας μαζί της θα ξεκινήσει 15 λεπτά αργότερα. Καλωσορίζω ε, μια ομάδα προσκεκλημένων του συναδέλφου Βίνκλερ, μέλη του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Σαξονίας από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ε, βρίσκονται στην αίθουσα ή δεν έχουν έρθει ακόμα οι προσκεκλημένοι του κυρίου Βίνκλερ. Εν πάση περιπτώσει τους καλυσορίζουμε και επειδή έχουμε καθυστερήσει να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια να μην ξεπεράσει τα πέντε λεπτά και μετά κάθε σκιώδη εισηγητή τρία λεπτά. Ελίζα Φερέιρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μην επαναλάβω στην προκειμένη περίπτωση αυτά που ήδη έχουμε συζητήσει και στην ε, υποβολή του σχεδίου Τη έκθεση στι 7 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα και θα προτιμούσα να επικεντρωθώ σε τρία-τέσσερα στοιχεία, σε τρια τεσσερα μηνύματα τα οποία έχω να σα απευθύνω. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπο με την εξή κατάσταση. Υπάρχει ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του πολίτη σε ό,τι αφορά τα θέματα τα φορολογικά. Το έχω πει και στο παρελθόν και το επιβεβαιώνω και τώρα. Το Κοινοβούλιο έχει και θεσμική ευθύνη. η οποία έχει να κάνει με την προβολή των φορολογικών ζητημάτων. Οι πολίτες προφανώς δεν είναι ικανοποιημένοι με την κατάσταση όπου η φορολογία πλήττει κυρίως τον πολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν ε, εστιάζεται ιδιαίτερα στις ε, πολυεθνικές εταιρείες. Ακόμα και οι χώρες οι οποίες απαιτούν από τους πολίτες ε, να κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες στα πλαίσια και του ευρώ, στις χώρες αυτές με την, με το ίδιο νόμισμα, με την ίδια εσωτερική αγορά, με την ίδια οικονομική πολιτική. Και στις χώρες λοιπόν αυτές υπάρχει το θέμα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Το θέμα λοιπόν είναι πολιτικό. Στο Κοινοβούλιο λοιπόν πλέον επαφίεται να αναλάβει δράση, να προβάλλει και να προωθήσει την ατζέντα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να συνεχίσει μία διαδικασία να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι και δίκαιο για τον πολίτη. Αυτό αποτελεί την ε, κορυφαία μας ευθύνη. Και θεωρώ ότι η μεγάλη και εντατική συνεργασία στο πλαίσιο του ανοιχτού χαρακτήρα και στο πλαίσιο της, ε, του συμβιβασμού και γι' αυτό ευχαριστώ τον ε, συνεισηγητή θα πετύχουμε αποτελέσματα. Η πρώτη μου λοιπόν έκκληση είναι να υποστηρίξουμε όλοι αυτό το βασικό μήνυμα που αποστέλουμε προκειμένου να καταλήξουμε όλοι σε έναν κοινό συμβιβασμό για να επιδείξουμε τη δέσμευση που έχουμε και να επιδείξουμε και προς το Συμβούλιο ποια είναι η στάση μας σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, τη δίκη διαμόρφωση της φορολογίας στην Ευρώπη. Κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω. το θέμα του θεσμικού, του θεσμικού σεβασμού των ε, δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Η ανταλλαγή πληροφοριών από τις πολυεθνικές εταιρείε είναι κάτι το ουσιώδες. Πολλές δεν έχουν ανταποκριθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη δική διαμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν πληροφορίες και από τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε πληροφορίες ε, τι τις οποίες ε, έχουμε ζητήσει και βάσει του κώδικα ε, δεν μα έχουν χορηγηθεί με την αιτιολογία της εμπιστευτικότητα. Έχουμε τα θέματα και τη Τραπεζική Ένωση. Στο παρελθόν υπήρχε το θέμα του απόρριτου το οποίο πλέον έχει ξεπεραστεί. Και αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι τα θέματα αυτά τα οποία αφορούν τόσο άμεσα τον πολίτη Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τέτοιες πληροφορίε να μην δημοσιοποιούνται στους εκπροσώπους. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση με την έγκριση του κειμένου όπως και ελπίζω, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω ό,τι αφορά την πολιτική πίεση που ασκούμε και όλα τα συνοδευτικά, όλες τις συνοδευτικές δράσεις για τα φορολογικά ζητήματα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες αρνήθηκαν να εμφανιστούν είναι γνωστές εταιρείε. Εταιρείε με κύρος, φήμη, η Amazon, ανέσαπος, Barclays Bank, η Coca-Cola, Facebook, Fiat, Chrysler, Google, HPC, IKEA, McDonald's, Philip Morris, Walmart, η Walt Disney Company. Και κάποιες από τις μεγάλες ε, εταιρείες ε, εμφανίστηκαν εδώ στο κοινοβούλιο, πήραν το λόγο. Η τάλ και άλλες εταιρείες, αυτές που ανέφεραν, αρνήθηκαν να χορηγήσουν τα στοιχεία αυτά. Πώς λοιπόν το Κοινοβούλιο γίνεται να επιδεικνύει τέτοιον ανοιχτό χαρακτήρα, ανοιχτό, ανοιχτό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη συζήτηση αυτή και να ζητάμε κανονικά από τις επιχειρήσεις να έρθουν κοντά μας και να μας ενημερώσουν. Επίσης, η Κομισιόν νομίζω πρέπει μάλλον να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στα κρατημέλη, ώστε να είναι ο κανόνας ο αμοιβαίος σεβασμός και εμείς μέσα σε αυστηρά όρια να συνεχίσουμε αυτή την εργασία. Γιατί διαφορετικά η πίεση η πολιτική ε, γίνεται διαρκής έτσι ώστε να επικρατήσει μια δικαιοσύνη στην εθνική αγορά, στην, στο ενιονόμισμα και βέβαια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ο Μίχαλ Τόιμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κοιτώντα ε, το, την απόσταση που έχουμε διανύσει, διαπιστώνουμε ότι υπήρχαν πολλά προσκόμματα. Ήταν ανηφορικός ο δρόμος παρά το γεγονός ότι εγκαίρως επισημάναμε στην έκθεση πρωτοβουλία και με τον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ ότι εκ των προτέρων δεν θα θέλαμε να επισκεφθούμε μόνο μία χώρα, όχι μόνο λοιπόν το Λουξεμβούργο, δεν ήταν το... στην αιστεία μόνο το Λουξεμβούργο, αλλά και άλλες χώρες. Είχα προτείνει λοιπόν εξ αρχής και την Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ελβετία, το Βέλγιο, ότι όλες αυτές τις χώρες λοιπόν έπρεπε να τις επισκεφθούμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και την εισηγητρία του στους συνεισηγητές για την μεγάλη απόσταση που έχουμε διανύσει, γιατί πραγματικά ήταν τεράστιο το πρόγραμμα εργασίας. Ε, πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις, διαπιστώσαμε και από τους ε, εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου ότι κάποιες χώρες έχουν ε, θέσει σε λειτουργία και έχουν εκμεταλλευτεί φορολογικά καθεστώτα για να ευνοούν τις επιχειρήσεις και πρόκειται για παραθυράκια. Αυτό είναι σαφές. Αλλά το βασικό ζήτημα δεν διευκρινίστηκε. Το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Αυτά τα παραθυράκια προέκυψαν ε, ως παράπλευρη απώλεια επειδή τα εθνικά φορολογικά σύστημα, συστήματα ε, και οι εθνικοί νομοθέτες τα έβλεπαν όλα από την εθνική προοπτική και έτσι κατάστρωσαν μία πολιτική, εθνική και το κίνδυνος και τα παραθυράκια προέκυψαν ως ε, παράπλευρη συνέπεια. και η οποία και αξιοποιήθηκε στη συνέχεια ως κατάσταση από τις διεθνείς ε, ε, και πολυεθνικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τις μεγάλες εταιρείε συμβουλευτική, με αποτέλεσμα μια μεγάλη Ιρλανδική εταιρεία να πληρώνει μηδενικό συντελεστή φορολογίας ή υπήρχαν πραγματικά στενές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων όπου θα πρέπει να θεωρήσουμε φυσικά ότι ήταν σκόπιμο σκόπιμη διαμόρφωση του συστήματος και η εκμετάλλευση του συστήματος. Αυτό δεν μπορέσαμε να το διευκρινίσουμε στις επισκέψεις μας επιτόπου. Γι' αυτό λοιπόν ε, περιμένουμε και απαντήσεις από τις συζητήσεις που συνεχίζουν να διεξαγάγονται. Και ελπίζουμε ότι και τα έγγραφα τα οποία που έχουμε ζητήσει θα τα λάβουμε. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν ζητήσει οι συνάδελφοι θα πρέπει να τα ξαναζητήσουμε και θα πρέπει να μας διευκρινίσουν τα άλλα θεσμικά όργανα κατά πόσο θα μας διαθέσουν αυτά τα έγγραφα. Δεν είναι δυνατόν τα θεσμικά όργανα και όλος ιδιαιτέρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέτει έγγραφα τα οποία δεν τα χορηγεί στους ερατούς εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα πώς θέλουμε να ασκήσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο ως θεσμικό όργανο αν δεν έχουμε τους πλήρεις φακέλους στους οποίους έχει δικαίωμα πρόσβαση στο Κοινοβουλίο. Γι' αυτό λοιπόν όπως είπαμε και στη συνεδρίαση των συντονιστών και επίσης όπως διευκρίνησε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να επιμείνουμε προκειμένου να λάβουμε τα στοιχεία αυτά. Και σε, περι... σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουν οι εργασίε τη Επιτροπής. Υπό όποια μορφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να αναβληθεί η έκθεση αυτή. Όχι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η έκθεση αυτή προκειμένου να διατηρηθεί και η ορμή που έχει δημιουργηθεί. Τώρα λοιπόν είναι η χρονική στιγμή και δεν θα πρέπει να αναβάλουμε την έκθεση. Και ένα τελευταίο στοιχείο για το πόσο αντιμετωπίζουμε τα πολυεθνικ... τις πολυεθνικές εταιρείες, τους πολυεθνικούς ομίλους. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ερετών εκπροσώπων του πολίτη το γεγονός ότι μεγάλη πολυεθνική όμιλη δεν δέχονται την πρόσκλησή μας να έρθουν στην Επιτροπή για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Αλλά οι λομπιίστες παράλληλα μας καλούν ως βουλευτές σε εκδηλώσεις όπου ε, το θέμα είναι η φορολογική, το φορολογικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα πρόσφατα έγινε και από την εταιρεία IKEA. Επαναλαμβάνω, εταιρείε που δεν έρχονται εδώ στην Επιτροπή μας να συζητήσουν και να λογοδοτήσουν, θα πρέπει να μπουν σε ένα μαύρο κατάλογο, σε μια μαύρη λίστα και να εξαιρεθούν από τις συζητήσεις και τη συμμετοχή εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Merci bien. Σας ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, μετά δηλαδή από όσα είπε ο εισηγητής, θα ήθελα να ε, σας ενημερώσω ότι μετά από την απόφαση που ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών πριν από δύο μέρες, έγραψα μια επιστολή την οποία θα λάβετε αντίγραφο ή έχετε ήδη λάβει αντίγραφο προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να ζητήσω τα διαπιστευτήρια των όσων έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο για τους εκπροσώπους των ε, επιχειρήσεων που δεν θέλησαν να απαντήσουν στην πρόσκλησή μας, συστηματικά να αποσύρονται, να ανακαλούνται. Πιστεύω λοιπόν πως το Κοινοβούλιο θα, μας, ε, θα δεχτεί το αίτημά μας. Επίσης εκφράσαμε την επιθυμία και να ε, επιστηθεί η προσοχή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων στην ανάγκη μέσα στο πλαίσιο της ε, τρέχουσας επαναδιαπραγμάτευσης των διοργανικών συμφωνιών ε, μεταξύ Κομισιών και ε, Κοινοβουλίου για την Μητρό των Ομάδων Πίεσης να προβλεφθούν κυρώσεις που δεν προβλέπονται πραγματικά μέχρι τώρα για τις περιπτώσεις όπου οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οργανισμών ή και μεμονωμένα άτομα τα οποία καλούνται να ε, εμφανιστούν ενώπιον ενός οργάνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόσκληση. Και φυσικά θα σας ενημερώσω για το ποια συνέχεια δόθηκε σε όλα αυτά. Και τώρα δίνω το λόγο στον σκιώδη συγκητή, και στην, δηλαδή στην Τανότα Χούμπνερ από το ΕΛΚΑ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω την πολιτική γραμμή που εξέφρασαν και οι δύο εισηγητές, αλλά και εσείς, Πρόεδρε, και να πω επίσης ότι πλησιάζουμε τη φάση όπου θα πρέπει να αξιολογήσουμε την σημασία του να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία ε, του σώματος για την εκθεσή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της εργασίας της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να εκφράσω, να αναφέρω μάλλον δύο-τρία σημαντικά θέματα που δεν κατάφερα να τα αναφέρω στην πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Τάξη και θα ήθελα να μιλήσω για τη διαφάνεια που είναι βασικό στοιχείο της αποστολής μας. Εδώ νομίζω όλοι συμφωνούμε. Ε, Επίση να πω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά πολύ ευφυής διαφάνεια, διότι θα πρέπει να δούμε ότι η διαφάνεια που προτείνουμε ε, θα προωθήσει την βελτιστοποίηση περαιτέρω. Και επίσης, επειδή δεν υπάρχει διάθεση για μεγάλη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της φορολόγησης, θα πρέπει να τα καταφέρουμε αλλιώς, μέσω μιας διαφάνειας. Ε, το, να καταφέρουμε δηλαδή μέσω της διαφάνειας τα όσα δεν καταφέρνουμε λόγω της έλλειψης ε, βούλησης για αναρμόνιση. Τώρα, για την αναχώρα έκθεση. Ε, το, ήθελα επίση να τονίσω την ανάγκη να μην υποτιμούμε το διοικητικό φόρτο που θα σήμαινε κάτι τέτοιο. Και δεν εννοώ μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις mid-caps που ελπίζω ότι θα εξερεθούν, αλλά να οργανώσουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, μπορέσουμε να καλύψουμε τις πολυεθνικές που είναι οργανωμένες ανά χώρα, παρότι έχουν πολλές θηγατρικές και υποκαταστήματα κτλ. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο νου μας όταν θα θεσπίσουμε τις προδιαγραφές για τις αναχώρα εκθέσεις και ε, έτσι να φροντίσουμε ώστε να μην είναι μόνο ένα κλικ στο πληκτρολόγιο, αλλά να προβλέπεται και επιπλέον αυτή η προσπάθεια για ε, την προσαρμογή των εταιριών. Τώρα, για τους ε, πληροφοριοδότες, η νομική, η παράνομη μάλλον συμπεριφορά πρέπει να αναφέρεται, αλλά πρέπει να αναφέρεται στις αρχές. Και στην περίπτωση όπου οι αρχές δεν αντιδράσουν, τότε θα πρέπει ο πληροφοριδότης να είναι προστατευόμενος και να μπορεί να απευθυνθεί και στο ευρύτερο κοινό. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που έχουμε πέρα από εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω ότι έχουμε και το θέμα της ε, ρύθμισης διαφορών. και να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε ένα σύστημα παγκόσμιας δεσμευτικής ε, διατησίας, αλλά και θέματα ε, διπλής φορολόγησης να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν έχει νόημα όλη αυτή η δήλωση γιατί πάρα πολλοί λομπίστες δεν θα συναντηθούν με τους ευρωβουλευτές ε, εκτός αν έχουν πρόσκληση ούτως ή άλλως οι περισσότεροι έτσι έρχονται να έχουμε name and shame να κατανομάσουμε δημόσια όλους αυτούς που δεν θέλησαν να συναντηθούν μαζί μας ή που δεν θα θελήσουν παρόλο που υπάρχει ο κίνδυνος να γελιοποιηθεί το ευαγές αυτό ίδρυμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να έχουμε μια θεσμική συζήτηση, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση στον κανονισμό να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο ε, ως συνέπεια κυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα, για την έκθεση. Δεν έχω πάρει απαντήσεις από τους δύο συνεισηγητές. Και μάλιστα για το βασικό ζήτημα. Τι είναι ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός. Όλοι λένε ότι ε, έχουν δικαίωμα να σχεδιάσουν το φορολογικό τους ε, καθεστώς, τις φορολογικές τους δράσεις, όπως σχεδιάζουν την ε, ζωή τους και στα υπόλοιπα σκέλη που τους αφαιρούν. Αυτό το παραδεχόμαστε όλοι. Τι σημαίνει όμως επιθετικότητα. Όλοι τι ξέρουμε όταν το βλέπουμε. πώ όμω το περιγράφουμε. Θέλω να είστε συγκεκριμένοι. Τι σημαίνει επιθετικό, φορολογικό σχεδιασμό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θυμάμαι με το LuxLeaks. Ποιο ήταν το βασικό ζήτημα. Και είχαμε και πολλές συζητήσεις με τον εισηγητή Τόιερ την ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, γιατί ως κράτος μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το φορολογικό σου σύστημα με τρόπο που θα ωφελήσει μια εταιρεία η οποία ανταγωνίζεται μια άλλη εταιρεία. Όπως και σαν κράτος δεν μπορείς να ενισχύσεις και να επιδοτήσεις μια συγκεκριμένη επιχείρηση που ανταγωνίζεται κάποια άλλη. Αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης και άρα ε, δεν, ε, και δυστυχώς δεν τονίζεται ιδιαίτερο στο σχέδιο έκθεσης. Γιατί οι συγητέ συμπεραίνουν ότι δεν διαπαραβιάζονται... ούτε υπάρχει δυνατότητα να παραβιαστούν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το μελετήσουμε πιο προσεκτικά αυτό. Και τέλος, επιδιώκω ή αδυνατό να αντιληφθώ τι κάνουμε με τις τρίτες χώρες, τις εξωτερικές δικαιοδοσίες τι θα εμποδίσει τις επιχειρήσεις που εδρεύουν τώρα στο Λουξεμβούργο να πάνε στο Λίχτενστάιν ή στις Ηνωμένε πολιτειε ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να έχει κανονισμούς που να ε, τις ευνοούν φορολογικά. Δεν είναι καλά συνταγμένα τα κεφάλαια ε, για αυτό το θέμα. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ συνάδελφε, αγαπητέ συνάδελφε, είναι πράγματι σημαντικές οι ερωτήσεις σας. Για την ΚΟΕ Φάμπιο Ντεμάση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι καταρχάς είναι η ώρα να πούμε μια αλήθεια που πονάει. Η αλήθεια που πονάει είναι ότι δεν μπορέσαμε να εκπληρώσουμε την εντολή μας. Όχι επειδή δεν θέλαν οι βουλευτές, αλλά επειδή η Κομισιόν, ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν μας διέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα. Ξέρω ε, ο κύριος Γιούγκερ και η κυρία Βέσσιγκερ ε, βγαίνουν και δηλώνουν ότι όλα έγιναν σωστά, αλλά εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις έχουμε ακούσει ήδη διαφορά σχόλια. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η εταιρεία ε, η εταιρεία IKEA να αρνείται να παραστεί εδώ πέρα στην Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και μετά να μας προσπαθεί να φάμε τα ωραία και φτεδάκια της. Είναι δικαίωμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε φυσικά την IKEA, αλλά αν κάποιος έρθει να ζητήσει, για παράδειγμα, επίσκεψη στην ε, πατρίδα μου, εγώ μπορώ να το διώξω έξω. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τους λομπιίστες να συνεχίσουν να προσπαθούν να... Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε τους λομπιίστες. Θα πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Μέστερ Σμιτ. Είμαι μειοψηφία βέβαια, αλλά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει επέκταση τη ε, εντολή τη Επιτροπή και να υπάρξει διερευνητική επιστολή. Το είχα πει εξ αρχή ότι υπήρχαν προβλήματα. Τώρα, για την έκθεση. Θα θέλαμε να υπήρχε λίγη παραπάνω τόλμη, για παράδειγμα, για τι συμβουλευτικέ ε, εταιρείε. Θα θέλαμε να αναφέρουμε με το όνομά του τις εταιρείε αυτές, η PricewaterCoopers, για παράδειγμα, και για του πολυεθνικού ομίλου. ισχύει το ίδιο. Η, Επιτροπή, η έκθεση επίσης αναφέρει αυτά που ανέφερε η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το CCCTB. Είναι σημαντικό εδώ να έχουμε έναν ε, τύπο που θα επικεντρώνεται στις ε, χρηματοπιστωτικές πτυχές και η ενοποίηση θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει στην, σε επιχειρήσεις να μετακινούν κεφάλαια ένθεν και ένθεν των συνόρων. Και ύστερα έχουμε και το θέμα της ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Πολλοί εμπειρογνώμονες από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο μας επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να είναι εντελώς διαφανής αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν αφορά αυτό επιχειρηματικά απόρριτα και θα συνεχίσουμε λοιπόν να ζητάμε να έχει το κοινό πρόσβαση εδώ, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε σωστή αντίδραση. Και οι εθνικοί νομοθέτες επέτρεψαν να εκμεταλλευτούν οι επιχειρήσεις την κατάσταση και στο country την ε, υποβολή αναφορών αναχώρα ισχύουν αντίστοιχα στοιχεία. Και εδώ συμφωνώ με την Τανούτα Μία επιπλέον κόκκινη γραμμή είναι να υπάρχουν ανώτατα όρια φορολογίες. Μα είναι δυνατόν μετά το LuxLeaks αυτό να είναι το συμπέρασμα τελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς πιστεύω ότι η Ελίζα Φερέιρα και ο Μίχαλ Τόιρ έδειξαν ότι υπάρχει τρόπος να συντάξει κανείς μια έκθεση με ουσιαστικές προτάσεις, άρα μια έκθεση φιλόδοξη, σε μια προσέγγιση ε, διακομματική θα το έλεγα. Τώρα θα πρέπει να διευρύνουμε αυτή την προσέγγιση και να απευθυνθούμε και σε άλλες πολιτικές ομάδες, ακολουθώντας το πνεύμα της ε, έκθεσης της Μαριάν Τάισεν στην προηγούμενη θητεία για τον εταιρικό φόρο. Υπάρχει τρόπος, είναι δυνατό. Η έκθεση έχει ουσία, έχει φιλοδοξία και ελπίζουμε να τύχει της πλειοψηφίας της έγκρισης, της έγκρισης της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας μιλήσουμε τώρα για τη διαδικασία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποδεχθούμε εδώ. Δεν χρειάζεται. Από τη στιγμή που υπήρξε τέτοια καθυστέρηση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποδεχθούμε και καλώς συντάξατε την επιστολή που συντάξατε. Τώρα, ως προς τα έγγραφα, δεν ζητήσαμε διερευνητική επιτροπή τυχαία. Το ζητήσαμε γιατί αυτή η επιτροπή έχει αρμοδιότητα πολύ πιο δεσμευτική έναντι των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Για συνένεση δεχθήκαμε η Επιτροπή αυτή να γίνει ειδική Επιτροπή και όχι Διερευνητική Επιτροπή. Άρα πρέπει εμείς να, να αρνηθούμε να μας ποδοπατήσουν και να μας περιφρονήσουν. Ορισμένα κράτη στο Συμβούλιο και τελικά ε, Πίσω από αυτή την περιφρόνηση ορισμένων κρατών μελών κρύβεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο χέρι μας είναι να μην το επιτρέψουμε αυτό. Υπάρχει καθυστέρηση, είναι σημαντικό να έχουμε φιλόδοξες προτάσεις και για τον ορισμό της ευθύνης και της αρμοδιότητας και για την διαδικασία και την κατανόηση των διαδικασιών μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις κλέβουν την εφορία ουσιαστικά. Αυτό είναι θέμα θεσμικής αξιοπρέπειας, αξιοπρέπειας των θεσμικών οργάνων και είναι θέμα που σχετίζεται άμεσα με την ικανότητά μας να εκπληρώσουμε το έργο μας, την αποστολή μας. Δεν πρέπει να επιδείξουμε αδυναμία και πρέπει να παρατείνουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας για τόσο χρόνο όσο δεν θα έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, δηλαδή μέχρι να την αποκτήσουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα αιτήματα ώστε από το καθεστώς όλο και μεγαλύτερης φορολογικής ανταγωνιστικότητας μεταξύ κρατών μελών να πάμε σε ένα καθεστώς περισσότερης συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και θα πρέπει να προστατεύσουμε και ε, τους whistleblowers, αυτός που ε, εγκαίρως ε, ε, σημαίνουν το καμπανάκι του συναγερμού, γιατί χάρη σε αυτούς τα μάθαμε και χωρίς αυτούς οι επιχειρήσεις θα συνέχισαν να ε, διάγουν έναν ήρεμο βίο και να πλέον σε καταγάλανα νερά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα μαζί. Μάρκο Τζάνι για το EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τη διαδικασία και εγώ επαναλαμβάνω πολύ γρήγορα κάποιες ε, έννοιες τις οποίες ήδη εξέφρασαν συνάδελφοι. Εμείς ως Επιτροπή, εμείς ως ε, μοναδικό θεσμό που εκλέγεται άμεσα από του πολίτε οφείλουμε να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε και να καταλάβουμε, να, να καταστήσουμε κατανοητό Ποιε είναι οι δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε εκτό των τυχών του θεσμικού μα οργάνου στην εκτέλεση της εντολής μας. Και είναι δυσκολίε που δεν προέρχονται μόνο από εξωτερικού παράγοντε, όπω οι πολυεθνικέ. Βεβαίω δεν μπορούμε να τι ξεχάσουμε. Ε, και, αλλά τι δυσκολίε που προέρχονται και από τα ίδια τα κράτη-μέλη και τα ε, θεσμούς της Ένωσης πολλές φορές ε, δεν μας επέτρεψαν να εκτελέσουμε την εντολή μας σωστά και με συγκεκριμένο σημείο. Αυτά όλα λοιπόν είναι καθήκον μας και είναι καθήκον μας γιατί ε, όλοι προσπαθήσαμε για αυτή τη δουλειά και οι πολίτες πιστεύουν στη δουλειά που κάνουμε. Ε, όσον αφορά τις πολυεθνικές, νομική βάση για να κάνουμε κάτι ε, έτσι, ε, έντονο ε, υπάρχει, αλλά μια έντονη δράση σημαίνει ότι θα πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι εμείς είμαστε ο, ο θεσμός, η Επιτροπή Τάξη κάνει μια σημαντική δουλειά και εσείς δεν μπορείτε να φέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο και να δείχνετε έλλειψη σεβασμού απέναντί μας. Ε, κάποιο τρόπο για να, δούμε, ε, για να δείξουμε ότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Είναι απαραίτητο όμως γι' αυτό να συμφωνήσουν οι περισσότεροι συνάδελφοι με αυτή την ε, προσέγγιση. Βέβαια, ε, για την ενδεχόμενη παράταση αυτής της εντολής είναι ε, αλήθεια ότι εμείς πρέπει να ε, τηρήσουμε μια προθεσμία και θα τη τηρήσουμε. Όμως, η δουλειά αυτής εδώ της Επιτροπής μπορεί και να συνεχιστεί. Μπορούμε να δώσουμε συνέχεια, μπορούμε να σκεφτούμε να προσθέσουμε κάτι σε αυτή την έκθεση, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για το περιεχόμενο το έχουμε ήδη συζητήσει, οπότε πολύ σύντομα θα σας πω ποιες θα είναι οι βασικές γραμμές για την ομάδα μου. Καταρχήν, και, για αυτή την, ε, και λόγω αυτής της συμπεριφοράς και αυτού του εμποδίου που συναντήσαμε από πλευράς των κρατών μελών και κάποιες φορές και από πλευράς της Κομισιόν και από την ομάδα του κώδικα διοντολογίας θα πρέπει να ενταχθεί κάποια σαφής αναφορά στην έκθεση αυτή όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες του. Γιατί δηλαδή συνέβη αυτό, γιατί συναντήσαμε δυσκολία στην εκτέλεση αυτή της εντολής και πιστεύω πως είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο σήμερα με τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον επίτροπο από Γιούνκερ να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Κατά τα λοιπά, προφανώς και θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε καλό συμβιβασμό ανάμεσα σε όλες τις ομάδες για να παρουσιάσουμε μια καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Θα έλεγα λοιπόν τώρα ότι τώρα όσον αφορά τα Υπουργεία Οικονομικών. Είχαμε στείλει επιστολή στην Προεδρία την, ε, του, του Λουξεμβούργου. Τότε ήταν η Λιθουανική. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαμε σε επαφή και με την ε, αυτή του Λουξεμβούργου. Και επίση σε όλου του υπουργού Οικονομικών των 28 κρατών μελών για το ε, περιεχόμενο της, της νομοθεσίας όσον αφορά τη φορολόγηση των εσόδων των επιχειρήσεων και μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ακόμα απαντήσει η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία και η Σλοβενία. Η Ιταλία μας απάντησε σήμερα το πρωί. Μετά, σύμφωνα με τα όσα μου ζήτησαν οι συντονιστές πριν δύο μέρες, εγώ παρενέβην Έκανα ε, διάβημα προς τους υπουργούς όλων αυτών των χωρών που είχαν καθυστερήσει. Η Ιταλία ανταποκρίθηκε και να θυμίσω ότι θα λάβουμε στις 22 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με αυτά που είχαμε προβλέψει πριν τις ε, διακοπές και χρειάστηκε να αναβάλουμε την, την συνεδρίασή μας λόγω της ελληνικής κρίσης τότε. Αλλά στις 22 λοιπόν Σεπτεμβρίου θα μπορέσουμε να ακροαστούμε τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου, προεδρεύοντα μάλλον του Συμβουλίου, τον τότε υπουργό του και νυν υπουργό του Λουξεμβούργου που θα μας ενημερώσει καθώς και τους τέσσερις υπουργούς Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Ελπίζω πως μέχρι τότε θα έχουμε και απαντήσεις από ε, χώρες που δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Γιατί διαφορετικά θα τους κατονομάσουμε. Και εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία αυτή τη συνεδρίαση που είναι δημόσια και αναμεταδίδεται στο ίντερνετ για να αρχίσω να το κάνω αυτό προφορικώς. Θέλετε κάτι ακόμα να πείτε Μάρτιν, κάποιο αστείο θέλετε μάλλον να μας πείτε. Βλέπω το πονηρό σας χαμόγελο. Μια σύντομη ερώτηση προς την πλειοψηφία της Επιτροπής εδώ που θα πρέπει να αποφασίσει. Γιατί έχουμε την αρχή της ισότητας εδώ. Οι ίδιες συνέπειες που, που αποφασίσαμε ε, ως πλειοψηφία για τις εταιρείες που δεν ανταποκρίθηκαν θα ισχύσουν και για τις κυβερνήσεις. Οι ίδιοι περιορισμοί θα ισχύσουν και για τις κυβερνήσεις να μας δώσουν πίσω τα, τις, τις κάρτες εισόδου τους. <laughs> για το ίδιο θέμα, Φιλίπ. Ναι. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Μέσερ Σμιτ, γιατί είναι χαρακτηριστική αυτή του η παρέμβαση. παρέμβαση ορισμένων πολιτικών ομάδων που βάζουν στι όρει τι δημοκρατίε και τι επιχειρήσει. Λε και ένα κράτο ήταν το ίδιο σαν μια εταιρεία. Κύριε Σμιτ, όσον με αφορά, είμαι καταρχήν δημοκράτη. και επειδή εγώ έχω εργαστεί 22 χρόνια σε μια ιδιωτική επιχείρηση, θεωρώ ότι οι επιχειρήσει είναι είναι υπηκόη κάθε δημοκρατίας και δεν ε, μπορούμε να τους θέτουμε στο ίδιο ε, βάθρο, στο ίδιο επίπεδο. Ναι, όμως έχει ένα... μια λογική σε αυτά που μας λέει ο κ. Μέσης γιατί έχουμε τη συμφωνία των συντονιστών ε, είχαμε συμφωνήσει να πάμε στη συνταγματική μας επιτροπή για το πρόβλημα των σχέσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα και στον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίρνει τα έγγραφα που χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών του το Κοινοβούλιο από τα άλλα όργανα και θα πρέπει να υπάρχει απλήρης διαφάνεια ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Προτείνω να σταματήσουμε εδώ τώρα αυτή την συναρπαστική συζήτηση όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ ε, κράτους και εταιρείας, αυτή τη φιλοσοφική συζήτηση. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν και στους υπολείπους. Ο κύριος Χάνεμανς από την ΕΝΕΦ. Όχι, δεν λείπει. Ο Φάβιο τώρα. Φάμπιο, είχατε ζητήσει να πείτε δύο λόγια για αυτή την αντιλαγή εδώ. Θα ήθελα να συστήσω στον κύριο Μέσσερ Σμιτ αν σκοπεύει να υποβάλει μια τέτοια τροπολογία σε ό,τι αφορά ε, την εξαίρεση και τον αποκλεισμό κάποιων κρατών μελών από τις Μεγάλες Βρετανίες θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Και πραγματικά θα ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω και το αποτέλεσμα. Ναι, αγαπητέ συνάδελφε, έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Τόιερ, αν μου επιτρέπετε. Όταν πήρατε το λόγο, μιλήσατε για τα κράτη-μέλη τα οποία μέσω της φορολογικής τους πολιτικής προσπαθούν να προσελκύσουν ορισμένες επιχειρήσεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να επικρίνουμε τέτοιου είδους προσπάθειες τόσο απλά. Άλλωστε, όλα αυτά εντάσσονται στην εθνική αρμοδιότητα. Το Λουξεμβούργο προσπαθεί να προσελκύσει επιχειρήσεις αλλά με εικονικό τρόπο. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν την έδρα τους εκεί, αλλά δεν έχουν εκεί την παραγωγή τους. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Από τα κράτη που πολύ απλά προσπαθούν να προσελκύσουν τις επιχειρήσεις και να έχουν εκεί πραγματική παραγωγή οι επιχειρήσεις αυτές. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμείς είμαστε υπέρ της αρχής σύμφωνα με την οποία οι φόροι πρέπει να πληρώνονται στη χώρα όπου ε, λαμβάνει η χώρα η παραγωγή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά. Πρώτα ο Μικαέλ να, να μας βγάλει τα συμπεράσματα αυτή της συζήτησης και μετά η Ελίζα. Μικαέλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να περιοριστώ στη μία ερώτηση η οποία μου τέθηκε άμεσα και να απαντήσω. Όντως, πρόκειται για ένα αποτελέσματα της Επιτροπής ότι οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι τα παραθυράκια αυτά λόγω της πολυσυνθετότητας των εθνικών νομοθεσιών προκύπτουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κατά πόσο είναι καλή ή κακή η εθνική νομοθεσία. Αν όμως δεν θέλουμε κάποιοι λίγοι ευρηματικοί, οι οποίοι έχουν και τα χρήματα να πληρώσουν τις ακριβές ε, εταιρείε συμβουλευτικής, ε, περιορίζουν στο μηδέν τους φόρους τους, ε, ενώ οι άλλοι που δεν έχουν τα χρήματα να τους πληρώσουν αυτούς τους συμβούλους επιχειρήσεων, τους φοροτεχνικούς, τελικά πληρώνουν φόρους. Πιστεύω ότι αυτό δεν αποτελεί δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό και εκεί εντοπίζω την ανάγκη ανάληψης δράσης. Τουλάχιστον και ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στην ιστορική αγορά, γιατί είναι διαφορετική κατάσταση από τον όσα. Γιατί στην ιστορική αγορά έχουμε την ελεύθερη μετακίνηση των κεφαλαίων και έτσι τα κράτη έχουν χάσει το δικαίωμα να φορολογούν στην πηγή του τα κέρδη. Αυτό προβλέπει η ελάχιστη φορολογική εναρμόνιση. Και γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με αυτά που προτείνουν οι συγητές. Merci, Elisa. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως ε, αυτή η συζήτηση ήταν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Αλλά το μεγάλο συμπέρασμα το οποίο αποκομίζω είναι ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία σύγκλησης ανάμεσα στη μεγάλη μετα... πλειοψηφία σχεδόν όλες τις ομάδες πολιτικές για αυτό το θέμα και γι' αυτό και η έκκλησή μου είναι ότι σεβόμενοι τις διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, να μπορέσουμε, ε, μπορέσαμε μάλλον να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Το κάναμε αυτό σε άλλες φάσεις, όπως με την έκθεση της, ήταν ένα παράδειγμα αυτής της ικανότητάς μας να συγκλίνουμε, έτσι ώστε το μήνυμα του Κοινοβουλίου ως ε, ενότης ε, οντότης που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιταχυνθεί και να κινηθεί το θεματολόγιο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο είναι υπό κατασκευή διαρκώς, δεν είναι κάτι το ολοκληρωμένο. Και είμαστε σε μια φάση όπου ακόμα μια φορά χρειάζεται μια νόθηση, ε, ακόμα μια, ένα λιθαράκι, ακόμα ένα πυλώνας, ακόμα ένα θεμέλιο σε, αυτή τη κοινή, ε, ε, σε αυτό το κοινό μας οικοδόμημα. Να μην πολλωθούμε ε, είναι είναι πολιτικός απαράδεκτο το κοινωνικό κόστος να βαραίνει τις μικρομεσαίες μόνο επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ε, γι' αυτό και είναι ένα θέμα σχετικής δικαιοσύνης. Άρα χωρίς σχετική δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Και γι' αυτό και ε, στο κοινοβούλιο, ε, το κοινοβούλιο βαραίνει αυτή η λειτουργία και από εμά εξαρτάται να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που χρειάζεται και να διαβιβάσουμε στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα την πολιτική όθηση που χρειάζεται για να μπορέσει να δοθεί η απαραίτητη όθεση. Και γι' αυτό και ανάμεσα στου δύο, δύο συντονιστές, δύο μάλλον συνεισηγητέ, παρά τι πολιτικέ μα διαφορέ, μπορέσαμε να βρούμε ε, συμφωνία, να βρούμε συνένεση για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση σε αυτό το τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κάτι που το χρειάζεται οπωσδήποτε και πηγόντω. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο να ζητά το λόγο σε αυτή τη φάση. Τέλεια. Οπότε σας προτείνω να διακόψουμε τις εργασίες μας και σας ζητώ να επανέλθετε όσο γίνεται πιο σύντομα μετά από την ψηφοφορία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ακρόαση όπως την επιθυμούμε. Διάλειμμα.